Colleagues, it's um, nine o'clock by... η ώρα είναι, βάσει του εντυχισμένου ορολογίου. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ίσως. Ξεκινώ με τις ανακοινώσεις του Προέδρου. σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρία των συντονιστών. Και έχουμε καταρχήν τον ορισμό των εισηγητών και εισηγητών γραμμοδότησης. Μια βασική έκθεση που αφορά τα ατυχήματα στην πολιτική αεροπορία. Το ΕΛΚ πήρε την έκθεση αυτή. Η κυρία Τιβέρακ είναι η συγγήτρια. Επίσης θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι εκ περιτροπής αναλαμβάνουν τις εκθέσεις οι ομάδες. Όσον αφορά τα πρότυπα εκπομπών αερίων σε σχέση με τα εμπορικά οχήματα τμήμα της ολοκληρωμένης στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τη μείωση των εκπομπών αερίων, γνωμοδότηση της ομάδας των ε, Ευρωπαίων ε, Συντηρητικών και όσον αφορά την γνωμοδότηση για την απαλλαγή, την ΕΜΣΑ, την ΕΑΣΑ, την ERA και την ΣΕΖ. Η ομάδα ALDE θα αναλάβει τις απαλλαγές αυτές. Επίσης λάβαμε κάποια έγγραφα ε, προς ενημέρωσή μας. In which the, uh, the... Οι εισηγητές θεώρησαν ότι δεν ε, χρειαζόταν ε, να γνωμοδοτήσουν. Επίσης όσον αφορά τον κανονισμό 2320 για τους κοινούς κανόνες ε, της, ε, πολιτικής, ε, της ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας. Μία ανακοίνωση που αφορά τις εσωτερικές διαστάσεις της ολοκληρωμένης θαλάσσιας στρατηγικής την εποπτεία, όπως επίσης και την έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, θαλάσσια στρατηγική, την ολοκληρωμένη. Δεν θα αναλυφθεί δράση εκεί, αλλά οι συντονιστέ ε, θεώρησαν ότι θα μπορούσε να είναι ένα τομέα όπου θα μπορούσαμε να, να ρωτήσουμε τον ε, υποψήφιο επίτροπο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι έχει νόημα αυτό. Επίσης, μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τη στρατηγική διεύρυνση και τις βασικές προκλήσεις 2009-2010. Ε, Οι συντονιστές προτείνουν ε, να μην υπάρξει τη γνωμοδότηση. Επίσης, ε, δεν θα αναλάβουμε δράση όσον αφορά την πρόταση για την ε, θέση σε σχέση με την τροποποίηση των παραρτημάτων 2 και 3 των πρωτοκόλων ε, της προστασίας της βιοπικιλότητας στη λεκάνη της Μεσογείου και αυτό είναι το 1 τρίτο του τίτλου που σας διάβασα. Αν θέλετε να διαβάσετε τον πλήρη τίτλο, μπορείτε να τον βρείτε στους φακέλους σας. Και επίσης, καμία δράση όσον αφορά την, ε, τα αλλιευτικά σκάφη, τη σχετική έκθεση όσον αφορά την ε, ιατρική θεραπεία εν πλώ. Επίσης αποφάσεις ε, όσον αφορά την, τις νομοδοτήσεις και τις ανακοινώσεις. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να πείτε? Όχι. Ωραία. Ακρόαση του υποψήφιου επιτρόπου για τις μεταφορές. Οι συντονιστέ αποφάσισαν ότι η ακρόαση σκοπό έχει να γίνει μια ζωηρή συζήτηση με τον υποψήφιο επίτροπο, μια ζωντανή συζήτηση και ότι πρέπει να αναφέρει τις πραγματικές του δεσμεύσεις ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών στο Κοινοβούλιο Όσον αφορά τι ενδεχόμενε ημερομηνίε, οι συντονιστές πρότειναν Ιανουάριο 2010, αντί, την ομα... αντί της εβδομάδας των Χριστουγέννων, που είναι μια φήμη που κυκλοφορεί στο Κοινοβούλιο. ότι μπορεί να κάνουμε ακροάσεις για τους επιτρόπους ε, την εβδομάδα που αρχίζει στις 21 Δεκεμβρίου. Εγώ είπα βέβαια στους ε, συντονιστές ότι ε, εγώ δεν μπορώ να, πάρω και διαζύγιο εκείνη την περίοδο. Δεν θέλω να το διακινδυνεύσω. Οπότε με ευγνώμων προς τους συντονιστές, επειδή προτίμησαν τελικά όχι το Δεκέμβριο, αλλά τον Ιανουάριο. Όσον αφορά την επιτροπολογία, Ο κύριος Καϊκόφ που, ήταν, ε, που είναι ο Διευθυντής ε, για την Εναέρια Ασφάλεια από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών ε, μας μίλησε για την πρόταση του Επιτρόπου Ταγιάννη όσον αφορά την μεταφορά υγρών στα αεροσκάφη. Την 1η Οκτωβρίου του 2009, του 2009 έγινε αυτό και έγινε και μία διεξοδική συζήτηση στους συντονιστές συμφωνήσαμε επί μίας πρότασης ε, δικής μου να καθοδηγήσουμε κάπως ε, την ε, συνεδρίωση των εθνικών εμπειρογνωμόνων που θα συνεδριάσουν για αυτό το θέμα κάποια στιγμή στο τέλος του τρέχοντος μηνός. Το πρώτο πράγμα που αποφασίσαμε είναι ότι ως πρώτο βήμα από το 2010 και μετά η μεταφορά υγρών θα επιτρέπονται σε ορισμένες σε συγκεκριμένες περιοχές ε, και υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Η πρώτη, το πρώτο αυτό βήμα θα βελτιώσει βέβαια την κατάσταση όσων έχουν αγοράσει κάτι από τα ε, καταστήματα των αεροδρομίων. Και η δεύτερη μας ε, απόφαση ήταν ότι μέχρι το 2012 όλες, ε, οι, όλα τα μηχανήματα, τα τύπου σε μηχανήματα, Μέχρι την, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2013 ε, σε όλα τα ε, αεροδρόμια που έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν όλα τα ε, υγρά βάση του κανονισμού 2028 Βέβαια δεν έχουμε τη δυνατότητα να γνωμοδοτήσουμε επισήμως. Ε, θα, πούμε και εμείς την τελική μας άποψη όταν η ομάδα των εμπειρογνωμόνων ε, θα έχει εκείνη γνωμοδοτήσει. Εμείς απλώς ε, είπαμε κάποιες προτάσεις ε, βάσει των οποίων θα μπορούσε να κινηθεί η Επιτροπή αυτή. Μάτια, θέλεις να σχολιάσω συγκεκριμένο θέμα? Είχαμε ακριβώς αυτή την ε, αίτηση να έχει κάποιος, να είναι κάποιος εκπρόσωπος από την Κομισιόν για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ναι, θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε καταρχήν ότι θα υπάρξει η διανομή του κειμένου σε όλους τους συναδέλφους, ώστε να είναι ενήμεροι για αυτό το κείμενο. Ε, αποζημίωση επιβατών αεροπορικών γραμμών σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρεία αυτής. Οι συντονιστές <clears throat> ε, θέσπισαν μια καταληκτική ημερομηνία μέχρι αύριο το μεσημέρι, ώστε το ψήφισμα αυτό να περάσει στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου, τη δεύτερη Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Εκεί λοιπόν θα ψηφιστεί αυτό το ψήφισμα μετά από τη συζήτηση που έχουμε διενεργήσει για τα προβλήματα που προκύπτουν από πτώχευση αεροπορικών εταιριών. Ακολουθεί το θέμα της διαλειτουργικότητος του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχέδιο προφορικής ερώτησης. Οι συντονιστές προτείνουν <clears throat> να υποβληθεί αυτή η προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου 2. Οπότε θα έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο θέματα μας για αυτή την Ολομέλεια. Στη συνέχεια, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις Γενικές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόεδρος της ε, Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών μου ζήτησε να αναθέσουμε σε ένα μέλος μας την ιδιαίτερη ευθύνη για όλα τα θέματα του mainstreaming, του gender mainstreaming. Και θα ζητήσω από την κυρία Τικάου να το πράξει αυτό. Αλλιώς ξέρω ότι και η κυρία Λίχτεμπερκ ενδιαφέρεται για αυτή τη θέση. Λοιπόν, με την άδειά σα ζητώ από την Αντιπρόεδρο κυρία Τικάου να αναλάβει αυτή την ε, ευθύνη, αυτή την αρμοδιότητα. Εάν δεν το θέλει, θα ζητήσω με την, ε, με την άδειά σα την κυρία Λίχτεμπεργκ. Ο κύριος, είχε, είχε κάνει μια πρόταση στη συνάντηση των συντονιστών, αλλά εγώ αρνήθηκα. Για τα διάφορα τώρα. συζητήσαμε το θέμα των εμπορευματικών διαδρόμων και οι συντονιστές τόνισαν κάποιες από τις δυσκολίες οι οποίες ανέκυψαν σε σχέση με το θέμα αυτό. Απλώς θέλαμε να τονίσουμε την ανάγκη να υπάρξει αγαστή συνεργασία μεταξύ του εισηγητή και των σκιωδών εισηγητών και ελπίζουμε τώρα ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί. <clears throat> Για την κλιματική αλλαγή, οι συντονιστές δέχτηκαν την πρόταση του κυρίου Αλ Καντράουι να έχουμε μια συζήτηση για τις μεταφορές και την κλιματική αλλαγή μαζί με την Κομισιόν στα πλαίσια της συνεδρίασης της Επιτροπής μας Μεταφορών πριν γίνει η συνδιάσκεψη Κοπενχάγης το Δεκέμβριο. Παρουσίαση μιας μελέτης για την Ευρωβινιέτα από το Κοινό Κέντρο Ερευνών και πάλι έγινε δεκτή πρόταση του κ. Ελ Καντράου από τους συντονιστές να προσκαλέσουμε το Κοινό Κέντρο Ερευνών για παρουσίαση και συζήτηση σε σχέση με την πρόσθετη μελέτη για την Ευρωβινιέτα, η οποία έχει ζητηθεί από το Συμβούλιο. Επίσκεψη στο ΕΜΖΕΡ. Έχουμε την πρόταση του κυρίου Ντερόιτερ, ο οποίος είναι ο εκτελεστικός διευθυντής του φορέου αυτού. Κάθε επιτροπή μπορεί να στείλει μια τριμελή αντιπροσωπεία στα, στους φορείς που είναι υπεύθυνοι για αυτούς, ο κύριος Στέξ και ο κύριος Βάνσεμ, που είναι οι υπεύθυνοι για τα θαλάσσια θέματα, θα πρέπει να πάνε, <clears throat> κατά την άποψή μου, στο ΕΜΖΕΡ. Και εγώ ή ο κύριος Ρίκη, ο αντιπρόεδρος, θα πάνε ως το τρίτο μέλος σε αυτή την αποστολή. Τέλος, ενημέρωση για την ε, πρωτοβουλία των Άλπαιων μεταξύ Αυστρίας και Ελβετίας για τη μεταφορά των αγαθών μέσω των Άλπων. Έχει προταθεί να γίνει μια άτυπη επίσκεψη στην Ελβετία στο τέλος της Ολομέλειας του Μαρτίου με στόχο να πληροφορηθούν τα μέλη της Επιτροπής μας και το προσωπικό σε σχέση με τη μεταφόρτωση αγαθών από οδικές σε σιδηροδρομικές μεταφορές. Οι πολιτικές ομάδες λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουν αν θέλει κάποιος να εκμεταλλευτεί αυτή την πρωτοβουλία. Αυτές είναι λοιπόν οι ανακοινώσει που ήθελα να σας κάνω σε σχέση με την ε, συνάντηση των συντονιστών. Κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ. Δεν θα σας διακόψω, Πρόεδρε. Εν τη ρήμη του λόγου σας. Σας ξέρω, σας ξέρω άλλωστε. Όσον αφορά την πρόταση ψηφίσματος, να επιστρέψουμε σε αυτό για την ε, πτώχευση των ε, αεροπορικών εταιριών. Δώσατε προθεσμία για αύριο για τι τροπολογίε και να ψηφιστεί την Ολομέλεια τη δεύτερη ή του Νοεμβρίου. Για τα σημεία 1 και 2. Μπορεί να κάνω λάθο, Λέει ότι έχει προβεί σε διαβουλεύσει, σε ευρείε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με του και έδωσε τα πορίσματα της μελέτης ε, στο Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Φεβράριο 2009 Πού βρίσκουμε αυτά τα πορίσματα, αν βοηθήσει κανείς. Εγώ δεν τα βρίσκω πουθενά. Πρόεδρος, θα προσπαθήσουμε να σας βρούμε μια απάντηση. Υποψιάζομαι ότι είναι στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν κάποιος από την γραμματεία μπορεί να βρει μια απάντηση που μπορούμε να βρούμε ένα αντίγραφο της εκθέσεως, θα σας ειδοποιήσουμε. Καλώς τίποτα άλλο όσον αφορά τους συντονιστές ιδεμή. Σας ευχαριστώ. Προχωρούμε. Στις διαθέσεις μεταφορές με σιδηρόδρομους, ε, διεθνών συνολικών μεταφορών, κοτίφ, στη σύμβαση αυτή. Ο κύριος, Κοτ, κύριος Κοχ θέλει να πει κάτι. Πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ντίτερ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το γεγονός ότι ακυρώνονται όλο και περισσότερες σιδηροδρομικές μεταφορές είναι κάτι το οποίο μας οδηγεί πολλές φορές σε οργή. Όλο και περισσότερα τέτοια επεισόδια έχουμε τα τελευταία χρόνια. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να καταλήξει σε μια συμφωνία για τη Διεθνή Συμφωνία Μεταφορών με Σιδηροδρόμο, την COTIF, η οποία υπάρχει ήδη από τη δεκαετία του 80 και όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσχωρήσει. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περισσότερο τι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες με τις όμορε χώρες. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προσχωρήσει πλήρω παρά το γεγονό ότι εκδήλωσε το ενδιαφέρον γιατί υπήρξαν νομικά προβλήματα στην υλοποίηση αυτή τη προσχώρηση. Τελικά λύθηκαν αυτά τα προβλήματα το Σεπτέμβριο και επομένω πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί πλέον να υλοποιήσει πλήρω αυτή την προσχώρησή τη στη συμφωνία. Επομένω, η θέση μα θα πρέπει να είναι θετική στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κόχ. Δεν ξέρω αν κάποιο από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει να σχολιάσει. Δεν είστε υποχρεωμένοι, αν δεν θέλετε. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ας δοκιμάσουμε χωρίς κάρτες, χωρίς ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αν έχουμε αμφιβολίες θα κάνουμε ηλεκτρονική. Ποιο είναι υπέρ, σηκώστε το χέρι παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Οπότε ομόφωνα. Συγχαρητήρια Ντίτερ. Θέλετε τους αριθμούς. Έχετε όλοι τις κάρτες σας για την ψηφοφορία ας το κάνουμε επίσημα, αριστοκρατικά, ηλεκτρονικά. Έχουμε, λείπουν δύο κάρτες αντιπροέδρων, να λέξουμε τις κάρτες. Γι' αυτό ήθελα να ψηφίσουμε το χέρι. Τέλος πάντων, ξεκινάμε την ψηφοφορία την ηλεκτρονική. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Ναι και Τέρμπιν, έχουμε 27 υπέρ, καμία κατά, καμία αποχή, 28, 29, προσθέτουμε, 30 υπέρ, έχουμε 30 υπέρ, καμία κατά, καμία αποχή. Ευχαριστώ κύριε Κόχ, συγχαρητήρια. Okay. Next. Πάμε παρακάτω. Να καλωσορίσω. Φτάσανε, μου φαίνεται. Καλωσορίζω λοιπόν στο Κοινοβούλιο μια ομάδα Καναδών βουλευτών και γερουσιαστών. Ο κύριος Μπράντμπορν, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για, την, για τη σχέση με τον Καναδά, έφερε αυτούς τους βουλευτές και ξέρω ότι θα γίνουν διάφορες συνεδριάσεις εργασίας και διακομματικές συνεδριάσεις για να αποκτήσουν μία άποψη για τις διάφορες στοιχές του κοινοβουλευτικού έργου όπως όταν έρχονται να μας ακούσουν εδώ, στην Επιτροπή μας. Σας εύχομαι λοιπόν καρποφόρες συζητήσεις εντός του Κοινοβουλίου και ευχάριστη διαμονή στις Βρυξέλλες. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Απευθύνω ένα καλωσόρισμα στους Καναδούς βουλευτές μας. Φιλοξενούμενους μας μάλλον. Μετά πάμε στο σημείο 9. ΕΦΗ e, συστήματα ποια είναι η κατάσταση. κυρία Γένσεν είναι η συγγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως τα θυμούνται τα μέλη της Επιτροπής τον Απρίλιο, το Κοινοβούλιο πριν τις εκλογές υιοθέτησε με μεγάλη πλειοψηφία την πρώτη ανάγνωση το θέμα αυτό των εφιών συστημάτων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εμπεριέχει σχέδιο δράσης για ευφυή e συστήματα μεταφορών και μία οδηγία πλαίσιο για ευφυή e συστήματα μεταφορών. Ποια είναι η ιδέα, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε να προωθήσουμε την χρήση ευφυών e συστημάτων μεταφορών στις οδικές μεταφορές και σε άλλους τρόπους μεταφορών, αλλά σε αυτή τη φάση κυρίως στις οδικές μεταφορές για να αυξήσουμε την ασφάλεια, την αποδοτικότητα στον αφορά τη χρήση ενεργείας και την αποτελεσματικότητα, την απόδοση, την καλή απόδοση των μεταφορών. Πολλά καλά απορρέουν από τα συστήματα μεταφορών, αλλά πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση όσον αφορά την χρήση αυτών των ευφυών συστημάτων. Και ίσως να χρειαστούν κάποιες προδιαγραφές, ούτω ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν ποιες προδιαγραφές πρέπει να εφαρμόσουν. Από πλευράς Κοινοβουλίου, επί Μακρόν, είχαμε συζητήσει το θέμα, έχουμε εκφράσει την άποψή μας και θα θυμόσαστε ότι τον Σεπτέμβριο η Επιτροπή Μεταφορών επιβεβαίωσε τη θέση του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση. Στο Συμβούλιο δεν υιοθετήθηκε ακόμα κάποιο κείμενο. Η Σουηδική Προεδρία εργάστηκε άοκνα πρόσφατα προσπαθώντας να αποφασιστεί μια θέση στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγώ και οι σκιώδεις εισηγητές συνεδριάσαμε δύο φορές με την Σουηδική Προεδρία καρποφόρες οι συζητήσεις. Σκοπός των συναντήσεων ήταν να εξετάσουμε τις 57 τροπολογίες του Κοινοβουλίου που αφορούσαν την οδηγία. Συζητήσαμε κάθε τροπολογία ξεχωριστά και ακούσαμε από πλευρά Συμβουλίου ποιες μπορούν να γίνουν αποδεκτές, ποιες όχι, που χρειάζεται κάποια διευκρίνηση. Και το θετικό της διαδικασίας ήταν ότι η θέση του Συμβουλίου συνέκλεινε με τη δική μας. Εξηγώντας τι θέλουμε να πετύχουμε μέσω των τροπολογιών μας, διευκολύνθηκε το έργο της Σουηδικής Προεδρίας να πείσει τα μέλη του Συμβουλίου ότι το να πλησιάσουν τις θέσεις μας ίσως θα ήταν καλή ιδέα. Αυτό που χρειάζομαι είναι να σιγουρευτώ ότι ανανεώνεται η εντολή που δίδεται σε μένα και στους κοιόδης εισηγητές αυτή που είχε, δηλαδή στα πλαίσια της συμφωνίας της πρώτης ανάγνωσης και θα ήθελα να ενημερώσω και την Επιτροπή σχετικά με το που βρισκόμαστε και προς τα που κατευθυνόμαστε. Και αυτό σύμφωνα με τον εσωτερικό μας κανονισμό. Έτσι πρέπει να κινηθούμε. Στόχος της Σουηδικής Προεδρίας είναι μια πρόορη δεύτερη ανάγνωση όπως αποκαλείται. Δηλαδή το Συμβούλιο να καταλήξει σε ένα κείμενο για την πρώτη του ανάγνωση, το οποίο θα μας βρίσκει συμφώνους και αυτό θα θεωρηθεί δεύτερη δική μας ανάγνωση. Δεν ξέρω αν θα συμβεί όμως αυτό. Όμως βλέπουμε μέχρι που μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα συναντηθούμε απόψε. Θα συζητήσουμε περισσότερα τεχνικά θέματα. Και σε τριμερή διάλογο θα προβούμε στο Στρασβούργο στις 24 ε, Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου θα σας ενημερώσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις κυρία Τσικάου, Βάιπολς ε, και τους άλλους για την επικοδομητική τους ε, συμμετοχή. Να συνοψίσω τον τριμερή διάλογο. Ακούστε και η θέση του Συμβουλίου για κάθε τροπολογία του Κοινοβουλίου. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιους τομείς έχουμε ίδια άποψη. Το Συμβούλιο συμφωνεί να εστιαστούμε σε, ε, σε προτεραιότητες υπηρεσιών και εφαρμογών. δεν δίνουμε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει προδιαγραφές σε όλους τους τομείς των έφιών συστημάτων, αλλά σε τέσσερις συγκεκριμένου. τομείς. τομείς. σε πραγματικό χρόνο για κυκλοφορία και ταξίδια, στοιχεία για ελεύθερες πληροφορίες καθολικές για την ε, συγκοινωνία, οικολογικά θέματα και ε, συστήματα κρατήσεων και θέσεις σταθμεύσεως ε, φορτηγών. Αυτοί είναι τέσσερις τομείς. Ίσως να μην συμφωνούμε ποια προτεραιότητα δίνουμε σε αυτούς τους τομείς, τους τέσσερις. Και περιορίσαμε το πεδίο για υιοθέτηση προδιαγραφών από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνούμε σε αυτό και το Συμβούλιο και εμεί. Συμφωνήσαμε στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και ή δυνατόν συμβατότητα των εφιών αυτών συστημάτων με παλαιότερα συστήματα. Δεν ήταν εύκολα. Ε, μα τα συζητήσουμε αυτά. Κάποια κράτη-μέλη ανησυχούσαν ιδιαίτερα. Και κάποιοι που γνωρίζει πολύ καλά ο πρόεδρος μάλλον, έχουν προχωρήσει αρκετά. Ίσως ανησυχίες για ήδη ε, χορηγηθήσεις επενδύσεις οδηγούν σε μεγάλους δισταγμούς, αλλά τελικά πλησιάζει η θέση του Συμβουλίου τη δική μας. Η συνέχεια των υπηρεσιών, το αδιάκοπο των υπηρεσιών αυτών, των ευφυών συστημάτων, αξιολόγηση συμμόρφωση και τυποποίηση και ε, διαλειτουργικότητα ήταν κάτι πάρα πολύ ε, σημαντικό για πολλά είδη μεταφορών. Έπρεπε να υπάρχει και σημείο διεπαφή με διάφορα άλλα είδη μεταφορών. Και συζητήσαμε και τους ευάλωτους χρήστε των μεταφορών, μια ορολογία που χρησιμοποιούμε στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στο κείμενο του Συμβουλίου, λέει ευάλωτοι χρήστε οδών και χρήστε με μειωμένη κινητικότητα. Πρέπει να συζητήσουμε την ορολογία, τι σημαίνουν αυτοί οι όροι και συμφωνούμε επί της διαδικασίας τροποποίησης προδιαγραφών και βασικών στοιχείων σε παραρτήματα ότι αυτά πρέπει να γίνουν μόνο της διαδικασίας συναποφάσεως. Δεν θέλουμε να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να αποφασίσει μόνη της. Αν πρέπει να αλλάξει κάτι θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο που δεν συμφωνούμε. Στον ορισμό του ελάχιστου επίπεδου για τα ευφύ συστήματα και το πώς ε, θα χρησιμο... σε τι επίπεδο θα χρησιμοποιηθούν. Υποχρεωτική χρήση. Αυτό είναι κάτι, η υποχρεωτική χρήση αυτών των συστημάτων είναι κάτι που φοβίζει τα κράτη-μέλη, φοβούνται ότι θα είναι κάτι πολύ δαπανηρό και δεν μπορούν να αποφασίσουν μόνο τους πότε θα μειωθεί το κόστος και είπανε με την οικονομική κρίση δεν μπορούμε να αφήσουμε εμείς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει πότε θα χρησιμοποιούνται αυτά τα συστήματα. Υπάρχει κάποιο περιθώριο, ίσως να εξετάσουμε αυτά τα θέματα ξανά και τις διαδικασίες για ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με, το, με το μέγεθος της κυκλοφορίας, κυκλοφοριακή συμφόρηση. Λοιπόν, υπάρχουν οι προδιαγραφές, όταν γίνει η χρήση και η εφαρμογή των συστημάτων, τότε ίσως τεθεί το θέμα των προδιαγραφών. Και επίσης είναι και το θέμα των ευθυνών, κάτι που τόνισαν οι εμπορευόμενοι, οι εμπλεκόμενοι. Εάν δεν επιληθεί το πρόβλημα των ευθυνών, τα ευφυή συστήματα δεν θα χρησιμοποιηθούν ευρύτερα αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Οι διατάξει περί προδιαγραφών για την προστασία των δεδομένων είναι άλλο πρόβλημα. Θέλουμε στο κείμενο να αναφέρεται ρητά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει δεν χρειάζεται, διότι έχουμε γενική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, δεν χρειάζεται μια ρητή μνήα σε αυτό το κείμενο. Όμω οι γενικοί κανόνε περί προστασία των δεδομένων δίνουν τη δυνατότητα δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένες διατάξεις σε μια συγκεκριμένη νομοθεσία. Και εδώ ε, χρησιμοποιούμε στοιχεία και επειδή ε, θέλουμε να προστατεύονται τα δεδομένα, θέλουμε να αναφέρεται ρητά αυτό το θέμα. Και αιτήσιος προγραμματισμός, και αυτό είναι κάτι που πρόκειται να συζητηθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε non-papers, έγγραφα εργασίες, για να εξηγήσει πώς θα γίνουν όλα αυτά και υποσχέθηκαν ένα νέο κείμενο για το θέμα των ευθυνών. Οπότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει σε όλη την διαδικασία. Συνοψίσαμε τα αποτελέσματα λοιπόν των δύο πρώτων τριμερών διαλόγων και οι πληροφορίες έχουν διαβιβαστεί και στους σκιώδεις εισηγητές. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να ανανεώσει την εντολή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων ή μπορείτε να μας πείτε τώρα, τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε πραγματικές διαπραγματεύσεις καλύπτοντας τα σημαντικά θέματα για το Κοινοβούλιο. Αυτά που προσπάθησα να σας περιγράψω και τα βασικά θέματα που είναι προς συζήτηση τα σημεία στα οποία διαφωνούμε. Το Συμβούλιο είναι υποχρεωτική χρήση αυτών των συστημάτων, το, οι διατάξει περί ευθυνών και οι διατάξει περί προστασία των δεδομένων. Υπάρχουν και άλλα θέματα, όπω ευάλωτοι χρήστε των μεταφορών, η λειτουργία τη συμβουλευτική ομάδα. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη των σκιωδών εισηγητών πάνω σε αυτά τα θέματα. Θέλω να πω ότι προσπάθησα να ακολουθήσω σφαιρική προσέγγιση. Από ό,τι καταλαβαίνω με τις νέες διαδικασίες, με τη συνθήκη της Λισαβόνα, ίσως να υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για το τι γίνεται και αν προχωράμε πολύ γρήγορα. Δεν είναι αυτή η δική μου πρόθεση. Πάντα είχαμε τη δυνατότητα να λέμε ότι δεν θέλουμε μια προώρη δεύτερη ανάγνωση αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Έχουμε όμως και μια ευκαιρία τώρα, διότι βλέπουμε ότι η Σουηδική Προεδρία χρησιμοποιεί αυτή τη διαδικασία του διαλόγου για να επηρεάσει τη συζητήση στο Συμβούλιο. Ήταν λοιπόν πολύ καρποφόρες οι συζητήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως μας πει κάτι για την υποχρεωτική ανάπτυξη αυτών των συστημάτων, τη χρήση τους. Ποιες είναι οι στο Συμβούλιο, το κόστος. Εγώ πάντα έλεγα ότι βεβαίω ίσως να χρειαστούν επενδύσεις που συνεπάγονται δαπάνες βέβαια αλλά γρήγορα θα υπάρξει ανάκτηση των επενδύσεων, απόσβεση των επενδύσεων και είναι μάλλον μικρές επενδύσεις σε σχέση με τις επενδύσεις που χρειάζονται για του δρόμου ή το ERTMS και άλλα συναφή συστήματα. Και στο τέλος θα ήθελα να πω ότι Ίσως θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη διάταξη περί επιτροπολογίας, κάτι που θα αλλάξει λόγω της συνθήκης της Και πρέπει να αλλάξει συνεπώς και το κείμενο. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως πάντα άλλαξε την ε, δομή του κειμένου. Αυτό μας δυσκολεύει τη ζωή θέλουν τα άρθρα να είναι λιγότερα, περισσότερες αιτιολογικές σκέψεις, περισσότερα στα παραρτήματα. Πρέπει αυτό να το εξετάσουμε όταν θα φτάσουμε στο τέλος. Δεν είναι ότι πρέπει να λάβουν πράγματα υπόψη, αλλά αν αυτά που περιγράφονται έχουν την ισχύ που επιθυμούμε εντό του κειμένου. Είναι και αυτό ένα θέμα που θα πρέπει να συζητήσουμε. Εάν θέλουμε να έχουμε μια πρόορη δεύτερη ανάγνωση, θα πρέπει να έχουμε ένα τελικό κείμενο στις 10 Δεκεμβρίου. Έχουμε συνάντηση Επιτροπής Μεταφορών 1η και 2 Δεκεμβρίου, οπότε έχουμε δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε το θέμα στην Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γένσεν, για όλα αυτά που μας είπατε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που εξακολουθούν ε, να υπάρχουν οι παλιές συνήθειες ε, ε, του τύπου «Αν έχετε αμφιβολίες, καλύτερα αιτιολογική σκέψη». Κύριο Κόχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω κυρία Γένσεν για την πολύ καλή πρότασή της. Εγώ νομίζω ότι καταρχήν είναι μια ενδιαφέρουσα προβληματική η οποία όμως περιέχει πολλές δυσκολίες. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εμπλεκομένων στο θέμα αυτό και θα ήθελα καταρχήν να εξασφαλίσω ότι θα ληφθεί υπόψη η άποψη όλων αυτών των εμπλεκομένων. Επί τη βάση του κειμένου της ε, Σουηδικής Προεδρίας δεν είναι δυνατόν να παίρνουμε το κείμενο χθε και να ψηφίσουμε σήμερα, να αποφασίζουμε σήμερα. Δεν είναι δυνατή λειτουργία αυτή μιας κοινοβουλευτική επιτροπή. <clears throat> Τώρα, Όλοι συμφωνούμε ότι τα ευφυή e e συστήματα μεταφορών είναι κάτι το θετικό, όπως τόνισε και η κυρία Γένσεν. Βέβαια, μέσα σε μια χρηματοοικονομική κρίση και η οικονομική κρίση είναι πολύ δύσκολο να επιβάλλουμε υποχρεωτικά την εφαρμογή τους. Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό όμως να δώσουμε δυνατότητα να έχουμε μια πιο αποδοτική σε σχέση με το κόστος μεταφορά, πιο φιλική προς το περιβάλλον και πιο καθαρή. Και αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα τμήμα των συγκυριακών προγραμμάτων τα οποία ε, θέτουν σε εφαρμογή τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσουν λοιπόν μέσω αυτών των προγραμμάτων να δημιουργήσουν μια καλύτερη οικονομική συγκυρία και όχι απλώς να αναμασίσουν τα προηγούμενα προγράμματα τα οποία είχαν χρησιμοποιήσει. Παραμένουν όμως πάρα πολλά να κάνουμε. Είναι ένας τρόπος για να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση στα ευφυή συστήματα μεταφορών και όχι για να δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα. Έχουμε επίσης το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Παρά το γεγονό ότι εγώ βλέπω ότι η κυρία Γένσεν προσπάθησε να το αντιμετωπίσει το θέμα αυτό πάρα πολύ επικοδομητικά. Αν δω το κείμενο όμω αυτό τη Προεδρία, όπου αλλάζουν τα πάντα, όπου το, οι αποφασιστικέ παράγραφοι γίνονται αιτιολογικές σκέψει, όπου αλλάζει η σειρά και, τον, και το περιεχόμενο των παραγράφων, όλα αυτά νομίζω ότι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό τρόπο, γιατί εμεί ως κοινοβούλιο δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι ουσιαστικό και τι δεν είναι ουσιαστικό, τι είναι αποδοτικό και τι δεν είναι. Θα ήθελα τώρα να σταθώ σε ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Παραδείγματο χάρη το e-call. Δεύτερον, τα θέματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων της αστικής ευθύνης και της διαλειτουργικότητας θα πρέπει να επιληθούν. Εάν αυτά δεν γίνουν, δεν υπάρξει σωστή διευκρίνησή τους και πάλι εγώ δεν μπορώ να ζητήσω από την πολιτική μου ομάδα να υπερψηφίσει στη δεύτερη ανάγνωση. Είναι απαραίτητο λοιπόν να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς λογικές, συμβιβαστικέ λύσεις για τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να διαπραγματευτούμε, αλλά δεν θα πρέπει να μας υποχρεώσουν με βεβαιασμένο τρόπο να καταλήξουμε σε μια απόφαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόχ. Ο κύριος Άλκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Τίκαου είναι η σκιώδη συζητήτρια, αλλά δεν μπορούσε να είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Συνεπώς, θα πω εγώ ορισμένα πράγματα εκ μέρους της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια γιατί μας έκανε μια πολύ καλή ενημέρωση και για την καλή συνεργασία που είχαμε μαζί της ως κοιόδης εισηγητές. Ε, το, τα ευφυή e συστήματα μεταφορών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο νομίζω ότι μπορεί να μας δώσει πολλές νέες δυνατότητες. Μπορεί να έχει ένα πολύ θετικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια, αλλά και στην αποτελεσματικότητα. και γενικώ ε, θα βοηθήσει πολύ την οργάνωση των μεταφορών μας. Ε, ακούστηκε το επιχείρημα, το επιχείρημα της οικονομικής κρίσης. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για τα επόμενα 10-20 χρόνια και ελπίζω ω τότε η οικονομική κρίση να έχει περάσει. Η άποψή μας είναι, σε γενικές γραμμές, ότι βεβαίως να σας υποστηρίξουμε, να προχωρήσουμε με τις διαπραγματεύσεις. Γνωρίζουμε ότι η θέση του Συμβουλίου απέχει αρκετά σε βασικά σημεία από τη δική μας και ελπίζουμε ότι μπορούμε να την προσεγγίσουμε και νομίζω επίσης ότι Τρία βασικά ζητήματα υπάρχουν. Πρώτον, υπάρχει το θέμα τη προστασία δεδομένων. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί στην οδηγία. Ε, το αναφέρατε και εσείς. Έχουμε, το θέμα της, ε, έχουμε την οδηγία προστασίας δεδομένων, αλλά χρειαζόμαστε πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές στο κείμενο, ώστε τα στοιχεία, τα δεδομένα να χρησιμοποιούνται σωστά και με ανώνυμο τρόπο. Ε, και επίσης ε, στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών ε, δεύτερη προτεραιότητα είναι το θέμα της ευθύνης και η σχετική ενημέρωση των εθνικών φορέων όπως επίσης και η υποχρεωτική ανάπτυξη των υπηρεσιών των εφιών συστημάτων. Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο, θα είναι δύσκολο να το συμφωνήσουμε και νομίζω ότι πρέπει να το διατηρήσουμε ως διαπραγματευτική θέση. Και για να ολοκληρώσω, η ομάδα μου εκφράζει την εμπιστοσύνη της ε, στην διαπραγματευτική ομάδα, στην εισηγήτρια και στους υπόλοιπους και όδης εισηγητές. Βέβαια πρέπει να δούμε και τα πιο λεπτομερή αποτελέσματα των ε, διαπραγματεύσεων. Στη συνέχεια, σε μεταγενέστερο στάδιο, και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, Στην επόμενη συνεδρία, σε αρχές Δεκεμβρίου, θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε μάλλον τα αποτελέσματα και να λάβουμε μια τελική απόφαση. Αλλά για την ώρα, βεβαίως, να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπρέπελς, από τους Πράσινους. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία <clears throat> εισηγήτρια, την κυρία Γένσεν, για τις εξηγήσει που μας έχει δώσει, οι οποίες ήταν πλήρεις και λεπτομεριακές σε σχέση με την κατάσταση των πραγμάτων. Επίση, για το γεγονός ότι πραγματικά έχει αναλάβει με πολύ ενεργητικό τρόπο αυτή την ε, προβληματική, αυτό το θέμα. Για το θέμα αυτό η ομάδα μου, οι πράσινοι, θεωρούν ότι οι διαδικασίες οι οποίες ε, προβλέπονται είναι ίσως ιδιαίτερα επαχθείς. Ο κύριος Κόκ ανέφερε ότι λάβαμε την τελευταία στιγμή το έγγραφο του Συμβουλίου και έχουμε την εντύπωση ότι έχει αλλάξει εκ το περιεχόμενο και η δομή αυτού του κειμένου. Ακόμα και χθε, που ήταν 9 Νοεμβρίου, είχαμε λάβει έγγραφα τα οποία είχαν ημερομηνία 30 Οκτωβρίου, δηλαδή πριν από 10 μέρες και επομένως θα πρέπει να δούμε κατά πόσο το Συμβούλιο πραγματικά ενδιαφέρεται να μπορέσει να εξασφαλίσει μια πρώιμη δεύτερη ανάγνωση. Εάν όμως πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να μας πάρει λίγο πιο σοβαρά το Συμβούλιο. Δεύτερον, το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης στάθμισε μια σαφή θέση σε σχέση με τα ευφύ συστήματα μεταφορών. Για μένα ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της πρώτης ανάγνωσης ήταν το εξής ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί κατά προτεραιότητα το σύστημα για την προστασία δεδομένων, της διαλειτουργικότητος και επίσης το θέμα των ευάλωτων χρηστών όπως και το θέμα της, του καταλογισμού της αστικής ευθύνης. Ένα σύνολο λοιπόν από ζητήματα, επίσης τα οποία εγώ δεν θέλω τώρα να τα απαριθμίσω, τα οποία όμως ενεκρίθησαν με μεγάλη πλειοψηφία από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπω εδώ τώρα ότι έχουμε από την πλευρά του Συμβουλίου μία θέση η οποία δεν ακολουθεί αυτά τα οποία ζήτησε το Κοινοβούλιο και ουσιαστικά η Κομισιόν σε αυτήν την περίπτωση συμπλέει με το Συμβούλιο. Εμείς λοιπόν δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο στόχος του Συμβουλίου στα πλαίσια αυτά. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα να αναφέρω τη δική μας θέση ότι η ομάδα μας είναι μεν απόλυτα διατεθειμένοι να διαπραγματευτούμε, να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμπεφωνημένο κείμενο μαζί με την συγγήτρια και τους υπόλοιπους συναδέλφους και να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια ταχεία δεύτερη ανάγνωση. Για μένα το πιο σημαντικό όμως είναι να μπορέσουν να διατηρηθούν τα κεκτημένα τη πρώτη ανάγνωση και να είναι το σημείο εκκίνηση περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φώστερ για το κόμμα των συντηρητικών. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ κύριε Πρόεδρε την κυρία Γένσεν για τις πλήρε εξηγήσει που έχει δώσει. Εγώ δεν γνωρίζω το θέμα αυτό, μόλις το αντιμετωπίζω και έχω ορισμένα ερωτήματα τα οποία χρήζουν διευκρίνησης, ίσως κάποιος από την Κομισιόν θα μπορούσε να απαντήσει, όχι τόσο κυρία Γένσεν. Μας λένε ότι στο μέλλον θα περιστοιχιζόμαστε από ευφύ συστήματα μεταφορών, είτε στον τομέα των ε, θαλασσίων μεταφορών, είτε των αεροπορικών, είτε των εμπαρευματικών μεταφορών. Αυτό για μένα είναι καλόδεκτο, είναι κάτι το οποίο φέρνει ήδη πολλά θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο ασφάλειας και σε άλλους τομείς για μας. Αλλά τα ερωτήματα τα οποία θέλω να θέσω και όπου ζητώ κάποια διευκρίνηση αναφέρονται περισσότερο στους οδηγούς, στους ε, γιοταχίδες. Πολλοί συνάδελφοι έχουν θέσει εδώ πέρα ορισμένα ζητήματα. Αν δούμε τι γίνεται σε επίπεδο κατασκευαστών αυτοκινήτων. Τι λέμε σε αυτό το έγγραφο. Λέμε ότι θα είναι υποχρεωτικό για όλα τα οχήματα, ανεξάρτητα από το αν είναι ακριβά και γεμάτα gadgets υψηλής τεχνολογίας, είτε είναι τα φθηνά αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί ο περισσότερο κόσμο. Θα πρέπει οι κατασκευαστέ αυτοκινήτων να βάζουν στα αυτοκίνητα υποχρεωτικά όλα αυτά τα μαύρα κουτιά που έχουν να κάνουν με τα ευφύ συστήματα. Είναι σωστό αυτό. Αυτό μας οδηγεί στο ερώτημα το οποίο έχει ήδη τεθεί για το πώς θα προστατεύεται η ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων. Κάθε φορά που μπαίνουμε στο αυτοκίνητό μας θα μας παρακολουθούν. Αν έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο, προφανώς ο καθένας ξέρει πού βρισκόμαστε. Αλλά το κινητό τηλέφωνο μπορούμε να το κλείσουμε. Με το αυτοκίνητο όμως, τι θα κάνουμε. Θα ήθελα λοιπόν να έχω περισσότερη εμπιστοσύνη σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους λοιπόν. Η τελευταία μου παρατήρηση επίσης είναι η εξής. Όταν προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την εναρμόνιση της τεχνολογίας, υπάρχει ελπίδα να καταλήξουμε σε κάποιο κοινό αποτέλεσμα, σε μια κοινή θέση. Αλλά υπάρχουν εταιρείε οι οποίε αναπτύσσουν τεχνολογία όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Ποιο θα αποφασίσει ποια είναι η τεχνολογία η οποία θα προκριθεί στον τομέα των ευφυών συστημάτων. Μπορεί κάποιε εταιρείε να έχουν ε, προωθήσει μεγάλες τεχνολογικές πρόοδους αλλά πώς αυτό το πράγμα θα ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια της εναρμόνισης. Για το θέμα αυτό λοιπόν θα ήθελα να έχω περισσότερες διευκρινήσεις από την πλευρά της Κομισιόν. Ο κύριος Μπραντβέρν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ έχω σοβαρέ ανησυχίε με την πρόταση αυτή, όπω και η κυρία Φώστερ. Αυτά τα νέα μαύρα κουτιά, όπω αναφέρονται στα μέσα μαζική ενημέρωση, και να είναι υποχρεωτικά σε όλα τα νέα οχήματα. Κοιτάξτε, όπως και η κυρία Γένσεν είπε στα εισαγωγικά της σχόλια, νομίζω ότι πηγαίνουμε πάλι προς ένα, μια κατάσταση εποπτείας και όπως είπε και η κυρία Φώστερ δικαίως, μπορούμε να δεχθούμε παρακολούθηση μέσω κινητών τηλεφώνων. Ήδη υπάρχει αυτό δηλαδή, αλλά δεν είναι δυνατόν να δίνουμε τη δυνατότητα ύπαρξης νέων συσκευών που όλο περισσότερο παρακολουθούν τον κόσμο. Καταλαβαίνω ότι οι προθέσεις είναι όσο το δυνατόν καλύτερες, αλλά πραγματικά δεν, χρειάζεται πολύ φαντασία για να καταλάβουμε πώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδου συσκευέ. και εγώ συνεπώς διαφωνώ με οποιαδήποτε υποχρεωτική εισαγωγή τέτοιου είδου τεχνολογία. Αυτό λοιπόν είναι το μειονέκτημα, κατά τη γνώμη μου. Τώρα, το, η καλή πλευρά που την ανέφερε και η κυρία Γένσεν στα σχόλιά τη είναι κάτι το οποίο μπορώ να καταλάβω και αφορά την ε, ασφαλή στάθμευση των φορτηγών. Είναι κάτι το οποίο δευρευνήσαμε πριν από 18 μήνες ε, και μάθαμε ότι υπάρχουν ε, κάποια σημεία στο Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον, στην πόλη μου για παράδειγμα, στο Μπέρμιγχαμ, υπήρχαν κάποια σημεία όπου υπήρχε ιδιαίτερη εγκληματικότητα κατά των φορτηγών και υπήρξαν κάποια πιλωτικά προγράμματα, για παράδειγμα στην νοτιοανατολική Αγγλία, ε, αλλά η πρόοδο ήταν πάρα πολύ αργή και γι' αυτό πρέπει να το εξετάσουμε με πολύ λεπτομέρεια το θέμα, να είναι ασφαλή, ασφαλής η χώρη στάθμευσης των φορτηγών να είναι διαθέσιμη και πρέπει να δούμε και πολιτικά πώς μπορούμε να το προωθήσουμε γιατί η εγκληματικότητα και οι απώλειες των φορτηγών είναι τεράστιες ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μορφή αυτή εγκληματικότητας και πρέπει να είναι μια προτεραιότητα την οποία πρέπει να την αντιμετωπίσουμε οπουδήποτε δεν είναι μόνο τεράστιες οικονομικές συνέπειες και καταστροφικές, αλλά προστατεύουμε τον κόσμο και τα αγαθά τους ε, κατά τις μεταφορές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπράντμπορν. Να πω και εγώ μερικά πράγματα σε σχέση με αυτό που είπατε και εγώ πιστεύω ότι αυτό το θέμα της ασφαλούς στάθμευσης των ε, φορτηγών είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Υπάρχει βέβαια πάντοτε ένα δίλημα. Όταν προτείνεται κάτι τέτοιο, όλοι οι ντόπιοι ε, δεν θέλουν να είναι κοντά στη πόλη τους ε, τα, οι χώροι αυτής στάθμευσης δεν, θέλουμε, δεν θέλει κανείς να είναι πολύ κοντά του τέτοιου είδους χώρη στάθμευσης, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να διερευνήσουμε αυτό το θέμα ε, της ε, ασφαλούς στάθμευσης των φορτηγών. Είναι πολύ σημαντικό. Και δύο κριτήρια υπάρχουν. Υπάρχει το θέμα της ασφάλειας το οποίο αναφερθήκατε και αν και υπάρχει και ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια. Γιατί υπάρχει και ένα θέμα οδική ασφάλεια όταν, αφορά, όταν ε, υπάρχουν χώροι ε, στάθμευσης των φορτηγών και σωστά ε, το αναφέρατε αυτό και νομίζω ότι το είπε και η κυρία Γένσεν στην παρουσίασή της. Αυτή η ασφαλής ε, στάθμευση των φορτηγών είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ιδιαίτερο πρόβλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος Στήλμαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πού είστε? Α, εκεί σας, είστε στο βάθος. Κύριε Τίλμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά της. Μας υποστηρίξατε πάρα πολύ ως Επιτροπή στην πρώτη ανάγνωση. Κάτι το οποίο νομίζω ότι συνεισέφερε πολύ στην ε, σημερινή κατάσταση. Πραγματικά το Συμβούλιο χρειάστηκε λίγο χρόνο για να, να φτάσει στο σημείο που είμαστε σήμερα. Αλλά και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μέσω τριμερών διαλόγων που έλαβαν χώρα πολύ πρόσφατα, με πολύ επικοδομητικό και ανοιχτό τρόπο, έδειξαν σαφέστατα τα προβλήματα που υπάρχουν για μια ενδεχόμενη συμφωνία. Επομένως, Πιστεύουμε ότι κατά τις επερχόμενες ημέρες και εβδομάδες θα γίνει σημαντική πρόοδος για την ε, ταχεία έγκριση του συγκεκριμένου εγγράφου. Και θα ήθελα να έρθω τώρα σε μερικά σχόλια που έκαναν ε, μέλη της Επιτροπής. Νομίζω ότι υπάρχει ευρεία ε, συνένεση όλων και του Συμβουλίου όσον αφορά τους στόχους και τη σημασία των ευφυών ε, συστημάτων μεταφορών για τις μεταφορές. Πραγματικά είναι μεγάλα τα ωφέλη αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και βεβαίως θα συνεισφέρει και στη μείωση των μοιραίων ατυχημάτων στον τομέα των ε, ε, μεταφορών. Δυστυχώς η Επιτροπή δεν ε, μπόρεσε ακόμη να προτείνει ευφυή συστήματα για όλα τα είδη μεταφορών. Βέβαια έχουμε λάβει υπόψη μας το σχετικό αίτημα του ε, Κοινοβουλίου και βεβαίως ε, θα το επεξεργαστούμε, αλλά είναι πολύ φιλόδοξο. Για την ώρα έχουμε αρκεστεί στη σύνδεση των οδικών μεταφορών με άλλα είδη μεταφορών, κάτι το οποίο πιστεύουμε ήδη ότι είναι φιλόδοξο και αν το δείτε και στη λεπτομέρειά του δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικότερα όταν μιλάμε για λεφτά. Οι επενδύσεις σε FEE e, συστήματα μεταφορών ε, χρειάζονται ιδιαίτερη υποδομή και είναι η υποδομή αυτή ε, κάτω του 10% με την, ε, με την εξαίρεση ενός 8%. Και βέβαια ε, το, το όφελος από τις επενδύσεις αυτές σε σχέση με την ασφάλεια είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχουν βέβαια κάποιες λεπτομέρειες που παραμένουν εκκρεμείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι υπάρχει και ένα ζήτημα προστασίας ε, και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Το ζήτημα λοιπόν αυτής ε, της, του ιδιωτικού βίου είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που για μας εξ αρχής ήταν πολύ σημαντικό. Είχαμε πει από την αρχή στην πρότασή μας ότι ε, είναι κάτι που πρέπει να γίνει σεβαστό και οτιδήποτε σχετικό υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Οδηγία το έχουμε λάβει υπόψη μας. Βεβαίω να βελτιώσουμε την κατάσταση για την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων, αλλά υπάρχει πάντοτε και το θέμα της ασφάλειας. Όταν μιλάμε για μια τομεακή οδηγία, για παράδειγμα τα FEE, συστήματα μεταφορών και αλλάξουμε τους γενικούς κανόνες, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ... Ε, να υπάρχει μια συνοχή. Δεν γίνεται να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου γενικοί κανόνες ε, ε, είναι εναρμονισμένοι, αλλά οι τομεακές οδηγίες δεν ακολουθούν. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιους ενδιασμούς ως προς την προσθήκη περισσότερων ε, στοιχείων για τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων, γιατί δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει η τομεακή οδηγία προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά την ευθύνη που είναι επίσης μια ανησυχία που ανέφεραν ε, μέλη της Επιτροπής. Η ευθύνη πρέπει να ορίζεται από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες Η στάθμευση των φορτηγών ε, που την αναφέρατε πολλές φορές. Να σας πω ένα παράδειγμα. 8 δισεκατομμύρια είναι η απώλεια ε, λόγω των ε, κλοπών που γίνονται σε φορτηγά κατά τη διάρκεια της στάθμευσής τους. Η ιδέα είναι να υπάρχει ένα σύστημα κράτηση των χώρων στάθμευσης από τους οδηγούς, ώστε να μπορούν να προγραμματίσουν το ταξίδι τους, να ε, βασίζονται στο γεγονός ότι θα, υπάρχει ένας χώρος στάθμευσης και να μην υπάρχει πρόβλημα όπως σήμερα που δεν υπάρχουν ε, ε, χώροι στάθμευσης συγκεκριμένοι, αρκετοί. υπάρχει πρόβλημα στάθμευσης, κάτι το οποίο δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο και για τα φορτηγά αλλά και για του ίδιου τους οδηγούς. Αν δεν βρουν θέση στάθμευσης, κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι επί του ζητήματος αυτού και πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα της ευθύνης που για την ώρα δεν το έχουμε σαφώς θέση στο πλαίσιο της οδηγίας. Όμως ευχαρίστως ε, να το επεξεργαστούμε. Ένα μεγάλο πρόβλημα μεταξύ ε, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου είναι η υποχρεωτική εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε όταν αποφασιστούν οι υπηρεσίες πρέπει να ε, αναπτυχθούν μετά. Διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα απλώς να ε, αποφασίζουμε για υπηρεσίες και ένα κράτος μέλος να τις εφαρμόζει άλλο όχι. Υπάρχει λοιπόν από τη μία το ελάχιστο οι ελάχιστες υπηρεσίες και οι χώροι στάθμευση ε, των φορτηγών που ανέφερα προηγουμένως ε, και αυτό θα έλεγα ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Είναι κάτι το οποίο επεσήμανε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση. Οπότε Ευχαρίστω να συνεργαστούμε και με το Συμβούλιο και με το Κοινοβούλιο για να βρούμε μια λύση για αυτή την υποχρεωτική ανάπτυξη υπηρεσιών. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ. Κυρία Γένσεν, θέλετε να πείτε τίποτα. Βασικά, οι συνάδελφοι είναι πολύ πρόθυμοι να σας δώσουν την εντολή και σε εσά και στους κοιόδης για να προχωρήσετε στις διαπραγματεύσεις. Δεν άκουσα αντίθετη άποψη. Άρα μπορείτε να προχωρήσετε από αυτή τη βάση. ώστε να πείτε τίποτα περισσότερο. Κυρία Γένσον, ευχαριστώ καταρχάς τους σκιώδεις για αυτά που είπαν. Yes, we got a text from, from council, but that has... Ναι, πήραμε το κείμενο από το Συμβούλιο, αλλά δεν είναι αυτό που συζητούσαμε. Συζητούσαμε τις δικές μας τροπολογίες. Εκεί βασιστήκαμε. Θέλαμε να δούμε χρησιμοποιώντας σαν αφετηρία τις δικές μας τροπολογίες μέχρι πού μπορούμε να προχωρήσουμε και πόσες θα δεχόταν το Συμβούλιο. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί βέβαια. Όταν θα εξετάζουμε το τελικό κείμενο. Έχει αλλάξει το κείμενο πάρα πολύ. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε το τελικό αποτέλεσμα βάσει του κειμένου. Αρκετοί αναφέρθηκαν στην ασφαλή στάθμευση των φορτηγών. Είναι ένα θέμα που το συζητήσαμε σοβαρά επί σειρά ετών στην Επιτροπή με τα δύο πιλωτικά προγράμματα. Ένα από αυτά εξακολουθεί και έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα για τους οδηγούς φορτηγών όπου μπορούν να κάνουν μια κράτηση για στάθμευση. Όλο και περισσότεροι ενδιαφέρονται και η Βελγική Προεδρία, η μελλοντική Βελγική Προεδρία μου είπε ότι θα συμπεριλάβουν αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη για να το εξετάσουν το θέμα τα κράτη-μέλη. Το μόνο που φοβάμαι είναι ότι ίσως να σκοτώσουν τον ιδιωτικό τομέα και να μην προβεί σε βήματα ο δημόσιος τομέας. Εμείς θέλουμε κάτι να γίνει για τους οδηγούς φορτηγών στην πράξη και όχι να καθόμαστε για να συζητάμε ποιο θα κάνει τι. Αυτό με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει ποιο θα βάλει το σύστημα, θέλω να υπάρχει. Εκεί πρέπει να εστιαστούμε στην Επιτροπή. Και γι' αυτό ε, χαίρομαι που συμπεριλαμβάνεται. Σαν τομέας όπου λέμε ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικός και νομίζω ότι θα πρέπει να εμείνουμε στις θέσεις μας όσον αφορά αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Κυρία Φώστερ, θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, σύντομα ερώτημα. Εγώ αναφέρθηκα στο μαύρο κουτί. Δηλαδή η τεχνολογία να μπαίνει υποχρεωτικά στα ταχύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μου διευκρινίσει περαιτέρω το θέμα. Κύριο κύριος Τίλμαν. Ναι, συγγνώμη, Λυσμόνησα αυτό το σημείο στην παρέμβασή μου. Δεν αφορά αυτό το μαύρο κουτί. Ας είμαστε ξεκάθαροι τα μαύρα κουτιά που δίνουν στοιχεία σε περίπτωση ατυχήματος σε αυτοκίνητο ή αεροσκάφος είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ δεν μιλάμε για μαύρα κουτιά σε αυτοκίνητα. Ναι, εντάξει, το καταλάβατε. Τα ακούσατε. Γιατί ήταν πολύ χαμηλόφωνη η εξήγηση. Καλώς. Όπως είπε ο στρατηγός Μακάρθουρ, θα επιστρέψουμε θα επιστρέψουμε στο θέμα στην επόμενη συνεδρίαση όταν ελπίζουμε ότι εσείς κυρία Γένσον θα έχετε να μας πείτε και άλλα πράγματα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία. Αυτό σημαίνει μόνο έναν άνθρωπο, έναν άντρα, τον κύριο Στέρξ, ο οποίος θα αναφέρει στο θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι, αν δεν σφάλω, πέρσι λοιπόν υπέβαλε μια πρόταση. Μάλλον αρχές αυτού του έτους. Μας έκανε μια πρόταση για μια ανακοίνωση και πρόταση οδηγίας. Στόχος τους για σύντομα ταξίδια των πλοίων να διευκολυνθούν οι διατυπώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ξέρω τι προσπαθούν να κάνουν και τους υποστηρίζω. Ας πάρουμε ένα φορτηγό που πάει από το Ροστόκ στη Βαλτική και θέλει να πάει στον Μπορντό. Να μπορεί να το κάνεις χωρίς να σταματήσεις πουθενά. Αν θες να κάνεις το ίδιο με ένα πλοίο, πρέπει να γεμίζεις έντυπα, παραέντυπα, κυρίως αν ξεκινήσει το πλοίο από την Αγία Πετρούπολη, που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μπαίνει σε ένα λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ενώσης και μετά συνεχίζει και πάει σε άλλο λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ενώσης με πολλά εμπορεύματα που θα παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε έχεις πολλά διοικητικά προβλήματα, γραφειοκρατία, χαρτούρα, οπότε η ναυσιπλοεία, που, η μεταφορά με πλοία που είναι φιλική προς το περιβάλλον είναι λιγότερο ανταγωνιστική διότι είναι πιο δύσκολο οι μεταφορές με πλοίο να ανταγωνιστούν τις οδικές μεταφορές. Άρα εγώ συμφωνώ απόλυτα με το σκοπό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχέδιο κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αποτέλεσμα εργασιών τριών γενικών διευθύνσεων. Αυτή, τις που ασχολείται με τα τελωνία, τις γενικές διευθύνσεις που ασχολείται με θέματα υγείας ας πούμε, έλεγχη επί εισαγωγμένων τροφίμων και η Γενική Διεύθυνση που ασχολείται με τις μεταφορές. Από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των τριών γενικών διευθύνσεων, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να σημειωθεί η πρόοδος. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστούν οι διευθύνσει μεταξύ του όσο γίνεται. Εάν δεν συνεργαστούν οι υπηρεσίε υγεία, τελωνίων και μεταφορών, ε, δεν θα τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να τονίσουμε. Δεύτερον, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται μια προσπάθεια για τυποποιημένα έντυπα που θα πρέπει να συμπληρώνονται και θα πρέπει να διατίθενται ηλεκτρονικά και θα μπορεί να γίνεται και η αποστολή των εντύπων ηλεκτρονικά και προς έκπληξή μου αυτό δεν ισχύει ακόμα σε πολλά λιμάνια και όλα αυτά τα συστήματα ανταλλαγής ηλεκτρονικών στοιχείων να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και να ενταχθούν σε ένα δίκτυο για τις ασφαλείς μεταφορές διαθαλάσσης. Είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται ήδη για τον έλεγχο των πλοίων, για τις ναυσιπλοείες των πλοίων, ούτω ώστε όσοι θέλουν να δουν τις πληροφορίες να μπορούν μέσω μιας ενιαίας θηρίδας, ενιαίου συστήματος να βρίσκουν τις πληροφορίες. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την ιδέα. Κρύβεται κάτι το οποίο υποστηρίζω πλήρως εγώ και ελπίζω και οι συνάδελφοι να υποστηρίξουν αυτή την ιδέα. Δηλαδή υπάρχει μια σύγχυση τώρα. Σύγχυση όσον αφορά την κατάσταση και είναι πολύ μεγάλη σύγχυση. Δεν μπορεί να μείνουν τα πράγματα όσο έχουν θα πρέπει να εξυγχρονιστεί το σύστημα. Και θα πρέπει ταχύτερο δυνατό να γίνει αυτό. Δεν θα επισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες, Πρόεδρε, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θέλω να υπογραμμίσω ως εισηγητής. Πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι η προθεσμία του 2010 να είναι πραγματική, τελική προθεσμία. Μου λένε ότι είναι τεχνικώς δύσκολο να προχωρήσουν πιο γρήγορα, αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα κράτη-μέλη καταλαβαίνουν ότι δεν πρέπει να κολλησιεργούν, διότι αν δεν λειτουργήσει το σύστημα μέχρι το 2013, μέχρι το 2010 διορθώνει ο μιλητής, θα έχουμε φύγει από την οικονομική κρίση και θα υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για τις μεταφορές. Οπότε ίσως να αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες αν δεν χρησιμοποιήσουμε όλους τους τρόπους μεταφορών και θα πρέπει να εφαρμοστεί η απλοποίηση μέχρι το 2010. Δηλαδή όλοι που συνδέονται με το ηλεκτρονικό σύστημα θα μπορούν να στέλνουν και να δέχονται αυτά τα έντυπα ηλεκτρονικά. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι δύσκολο και για το οποίο δεν έχει θέση χρονοδιάγραμμα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι κάτι που απαιτεί από τα κράτη-μέλη. Είναι το γλωσσικό θέμα, η γλώσσα. Προφανώς αυτό είναι ένα θέμα που δημιουργεί πάντα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν υπάρχει κάποια άποψη για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Να αφήσουμε όλους να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους, αυτό που συμβαίνει τώρα, αλλά δημιουργεί προβλήματα. Θα πρέπει να περιοριστούμε στις γλώσσες εκείνες που χρησιμοποιούνται στον IMO και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τρεις γλώσσες βασικά, ή θα πρέπει να προτείνουμε όπως και στις αερομεταφορές να χρησιμοποιούνται τα αγγλικά. Τα είναι η γλώσσα επικοινωνίας η αγγλική. Η δική μου άποψη, δεν ξέρω ποια είναι το συναδέλφων, δική μου άποψη είναι να ζητήσουμε να απλουστευτεί στο βαθμό του δυνατού η διαδικασία και να κάνουμε αυτό που γίνεται σε πολλά μέρη στην πράξη. Δηλαδή να χρησιμοποιείται η αγγλική σαν κοινή δεύτερη γλώσσα. Θα ήθελα να περασπιστώ αυτή την ιδέα, Πρόεδρε. Ξέρω ότι είναι ευαίσθητο θέμα, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο για τις θαλάσσιες μεταφορές να προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε αυτή την πτυχή στην πρότασή μας. Κάτι που ήδη εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις στην πράξη. Κάτι άλλο που δεν θεωρεί τόσο κατεπήγον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάνει κάποια σύσταση προς τα κάτι μέλη είναι και το εξή. Οι υπηρεσίες πλοήγησης και οι υπηρεσίες, η πληρωμή των υπηρεσιών. Όταν μπαίνει ένα πλοίο σε ένα λιμάνι, πολύ συχνά είναι καλό ο πλοίαρχος να έχει και πιστοποιητικό πλοήγησης για το συγκεκριμένο λιμάνι υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Το χρησιμοποιούν αυτό σαν δικαιολογία τα κρατη για να προστατεύουν τους πλοηγούς ε, με το επιχείρημα της ασφάλειας. Αλλά μπορεί ο καπετάνιος που επισκέπτεται συχνά ένα λιμάνι να ξέρει καλά τις δεπτομέρειες του λιμανιού και να κάνει τη δουλειά του πλοηγού και να έχει ένα πιστοποιητικό εξαίρεσης από παροχή υπηρεσιών πλοήγησης. Θα πρέπει λοιπόν να χορηγούνται αυτά τα πιστοποιητικά, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να είναι συγκρίσιμη η πρακτική αυτή που θα ακολουθείτε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξέρει ο τομέα ποιε είναι οι απαιτήσει και αυτέ οι απαιτήσει να είναι αναλογικέ. Δεν μπορεί κανεί να επιβάλλει δυσανάλογε απαιτήσει που να έχουν προστατευτικό χαρακτήρα. Θα πρέπει να, οι απαιτήσει να έχουν το στοιχείο τη αναλογία. Γνωρίζω ότι μιλάμε για ασφάλεια και δεν μπορούμε να κάνουμε παραχωρήσει σε θέματα ασφαλείας, αλλά νομίζω ότι για τα σύντομα αυτά, σύντομες διαδρομές της θαλάσσιας, να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι πρακτικά και να κάνουμε την αυσιπλοή αυτή μικρών αποστάσεων βιώσιμη. Θα πρέπει να εξετάσουμε και τη δυνατότητα ενθαρρύνσεως των διαφόρων ώστε να μην συμπεραβάνουμε μόνο τα θαλάσσια λιμάνια, αλλά να εξετάσουμε και τα ζητήματα εσωτερική ναυσιπλοεία. Να καλύπτει και εσωτερική ναυσιπλοεία. Η απλούστευση των κανόνων δεν πρέπει να σταματάει στα θαλάσσια λιμάνια. Μπορούμε να προχωρήσουμε και πιο πέρα, να κάνουμε άλλο ένα βήμα. Και αν έχουμε κόμβου εσωτερική ναυσιπλοεία που μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα, τότε μπορεί να προχωρήσει ακόμα ένα βήμα η απλούστευση. Να εξεταστεί δηλαδή ο συνδυασμό θαλάσσιας ναυσιπλοείας και εσωτερικής ναυσιπλοείας και αυτά να συνδεθούν μεταξύ τους, να συνδεθούν τα συστήματα αυτά μεταφορών, θαλασσίων μεταφορών και εσωτερικής ναυσιπλοείας και να καλυφθούν από αυτή την απλούστευση. Όσο μπορούμε να προχωρήσουμε όσον αφορά την απλούστευση, καλό θα είναι. Και σίγουρα είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτό το δίκτυο που δημιουργήσουμε θα είναι, ένα, θα είναι μια ενιαία θηρίδα που μπορεί να βρει κανεί όλε τι πληροφορίε αυτό το δίκτυο για την ασφαλή ναυσιπλοεία, θαλάσσια ναυσιπλοεία. Τώρα, όσον αφορά τον έλεγχο τη ναυσιπλοεία, είναι κάτι που βασίζεται στη συνθήκη τη Λισαβόνα. Θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερε πληροφορίε που διατίθενται για τα εμπορεύματα, για το φορτίο, Πληροφορίε που χρησιμοποιούνται από τι τελωνιακέ υπηρεσίε και από άλλε υπηρεσίε επίση. Χρειαζόμαστε αναβάθμιση του υφισταμένου συστήματο, ούτω ώστε να υπάρχει επαφή μεταξύ των διαφόρων υπευθύνων. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτού του υπεύθυνου να ανταλλάσσουν τι πληροφορίε, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το προωθήσει αυτό. Αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα, e-customs, το ηλεκτρονικό σύστημα τελωνίων θα πρέπει να καλύπτεται, να μπει, να ενταχθεί στο δίκτυο. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό, και το συζήτησα με του ανθρώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λένε ότι είναι σημαντικό να προσθέσει κάτι το Κοινοβούλιο. Ποιο είναι το σημαντικό, πρόσβαση στι πληροφορίε είναι σημαντικό στοιχείο. Προφανώ κάποιε από τι πληροφορίε θα πρέπει να είναι προσβάσιμε για ευρύτερο κοινό, αλλά αν πρόκειται να ανταλλαγούν πληροφορίε περί φορτίου που μεταφέρεται από κάποιο πλοίο, τότε η πρόσβαση πρέπει να είναι περιορισμένη σε εκείνου που χρειάζονται τι πληροφορίε. Θα πρέπει να καθορίσουμε σαφώς Ποιο έχει πρόσβαση στι πληροφορίε αυτέ, ποιο τι χρειάζεται αυτές τις πληροφορίες, διότι ίσω να μιλάμε για πολύ ευαίσθητε εμπορικέ πληροφορίε. Ένα πλοίο με έναν πλειοκτήτη που δεν θέλει οι ανταγωνιστές του να έχουν όλες τις πληροφορίες για το πλήρωμά του, για τα φορτία που μεταφέρει και ούτω καθεξής. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, Πρόεδρε, Πιστεύω το Κοινοβούλιο πρέπει να επιμείνει για την ταχύτερη δυνατή διεκπαιρέωση του ζητήματος και θα πρέπει να τηρήσουμε την προθεσμία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2013 και στις διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο θα πρέπει να παραμείνουμε σε αυτή τη θέση. Αυτά έχω να πω. Περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω τις σκέψεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στέρξ. Τη στιγμή που τα αγγλικά είναι η δεύτερη μου γλώσσα, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η πρότασή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα αγγλικά σαν μια κοινή γλώσσα. Κύριε Πασκουά από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινούμε σήμερα την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την πρόταση οδηγία της το, τις, για τα θέματα ναυσιπλοίας. Ο κύριος Στέρξ, ο συγητής, έχει παρουσιάσει τις γενικές κατευθυντήρες γραμμές της έκθεσής του και νομίζω ότι δεν θα έχουμε δυσκολία να συμφωνήσουμε μαζί του. Είναι απαραίτητο η κοινή λογική να πριτανεύσει ή να υπάρξει μια αντιμετώπιση ορθολογισμού και αποτελεσματικότητας. Νομίζω λοιπόν θα μπορέσουμε να βρούμε κοινέ λύσεις μαζί με τον κύριο Στέρξ. Αυτό το εγχείρημα έχει να κάνει με την συνολική προσπάθεια για μια διαλειτουργικότητα. Να μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε μια σωστή σύνδεση όλων των ε, μέσων των θαλασσίων και εσωτερικών υδατίνων δρόμων ε, στα μέσα μεταφοράς. Πολλές φορές έχουμε πάντα προβλήματα με τους ε, νομομαθείς, με εξωτερικούς φορείς που μας λένε ότι όλα αυτά είναι πρόωρα, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα, ότι πρέπει να περιμένουμε να συσσωρεύσουμε τις απαραίτητες εμπειρίες. Εγώ όμως πιστεύω το αντίθετο, ότι δεν πρέπει να αναμείνουμε. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πρωτοπόρο στον τομέα αυτό και να πρέπει να προωθήσει το θέμα αυτό. Η πρόταση οδηγία λοιπόν νομίζω αυτό το οποίο προσπαθεί να επιτύχει είναι να μειώσει και να απλοποιήσει τους ελέγχους είτε ουσιαστικούς ελέγχους είτε ελέγχους εγγράφων για τα πλοία και τα εμπορεύοντα που μετακινούνται μεταξύ των λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό ενιαίο χώρο θαλασσίων μεταφορών χωρίς κανένα φραγμό. Ένα ακόμα όνειρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης να ευνοήσει τις μεταφορές βραχαίων διαστα... Ε, αποστάσεων για να μπορέσει επομένω να ευνοήσει ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να παίζει ένα πρωτοπόρο ρόλο σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση του διεθνούς δικαίου και των συμβάσεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στην ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί που λένε ότι δεν πρέπει να κινούμεθα με ταχεία, ταχεία βήματα, πρέπει απλώ να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι άλλοι. Όχι, λέω, η Ευρώπη θα πρέπει να προωθήσει τον εξυγχρονισμό. Θα πρέπει <clears throat> να ενσωματώσουμε λοιπόν συμβάσεις όπως σύμβαση ΦΑΛ χρειάζεται να εξυγχρονίσουμε το σύστημα πληροφοριών, το SafeCNet, SafetyNet. Να μπορέσουμε λοιπόν το SafeCNet να ενσωματώσουμε λοιπόν το σύστημα πληροφοριών θα ευνοήσει ιδιαίτερα την ασφάλεια στο θαλάσσιο χώρο. Λέω και πάλι ότι όπως και ο κύριος Στέρξ υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει να χρονοτριβήσουμε, θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την γραμμή της Κομισιόν χωρίς καμία χρονοτριβή και τέλος η πρόταση αυτή για μένα είναι πάρα πολύ θετική. Μπορούμε να συζητήσουμε επί των λεπτομεριών. Θα έχουμε τον απαραίτητο χρόνο να το κάνουμε αυτό. Α, θα πρέπει να αναμείνουμε την πρόταση του κύριου Στέρξ, στην οποία πιστεύω ότι θα επικρατήσει η σωστή λογική του κυρίου Στέρξ και για μένα είναι θεμελιώδες για την ανάπτυξη της, ε, των θαλασσίων μεταφορών βραχαίων αποστάσεων να κάνουμε όλα αυτά τα μέτρα, γιατί αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ναυσιπλοεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιλάνα. Κοιτάξτε, δεν ξέρω πολύ καλά τον κύριο Στέρεξ, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο τρόπος, ο, η ανάλυση που έκανε, η παρουσίαση που έκανε, δείχνουν ότι μπορούμε να κάνουμε άριστη κοινή δουλειά ε, και με μένα και με τους άλλους σκιώδεις μπορούμε να κάνουμε καλή δουλειά μαζί. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό όσον αφορά τη αστηριότητα και εγώ έχω εμπιστοσύνη σε όσα είπε ο συνάδελφος και όπως τοποθετηθήκε. Από πρώτη ματιά αυτή η ανακοίνωση φαίνεται να είναι κάτι εξαιρετικά τεχνικό ασχολείται με αυτή και άλλες δράσεις του τομέα αυτού που έχουν στόχο να εγγυηθούν την επέκταση της αγοράς, εσωτερικής αγοράς θαλασσίων μεταφορών. Θα κάνουμε λάθος αν η προσέγγιση μας είναι απλώς τεχνικής φύσεως. Θα πρέπει να πεσιώσουμε τη δράση μας σε ανανεωμένη ανταγωνιστικότητα που μπορεί να έχει το τομέα θαλασσίων μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να οικοδομήσουμε έτσι ε, μία άλλη φάση αναπτύξεως θα πρέπει να ακουστούν απόψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περνάμε φάση ανταλλαγή απόψεων και θα πρέπει να προχωρήσουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να είναι μια πρώτη, ε, πρώτο βήμα απλούστευση που θα ε, οδηγήσει σε ανταγωνιστικότητα των θαλασσίων μεταφορών εν συγκρίση με τις χεσές μεταφορές. Λοιπόν, αν συμφωνούμε όλοι. Εγώ θα έδινα μεγάλη προσοχή σε αυτή την τοποθέτηση. Συμφωνώ ότι πράγματι ότι το χρονοδιάγραμμα, ο χρονισμός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται, αν υπάρχει περιθώριο να επιταχύνουμε κατά λοιπά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν πιεστεί, να προχωρήσουμε πιο γρήγορα θα πρέπει να βρούμε απαντήσεις συγκεκριμένα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Διαπλές ε, προτάσεις σε αυτή τη φάση για να συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες εβδομάδες. Εγώ θα έκανα διάκριση μεταξύ των δύο βασικών θεμάτων. Πρώτα απ' όλα έχουμε την πτυχή της απλούστευσης της χαρτούρας, ούτως υπήν, δηλαδή τα επίπεδα τεκμηρίωσης που απαιτούνται και έχουμε μια πτυχή γραφειοκρατική που θα πρέπει να απλουστευτεί όσον αφορά τι εσωτερικέ μεταφορέ Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Δεύτερο στοιχείο. Και εδώ ίσως η ανακοίνωση μπορεί να εμβαθύνει περισσότερο. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο θάρρος, θα έλεγα. Πρέπει να δούμε τι γίνεται σε εσές μεταφορές. Τα λιμάνια μας είναι διαφορετικά. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα ε, επιμελητίας πολλές φορές όταν φτάνει ένα πλοίο δεν βρίσκει την κατάλληλη, τα κατάλληλα μέσα, την κατάλληλη εξυπηρέτηση. Ε, θα πρέπει να δούμε πώς η, ο εκτελονισμός, όταν φτάνει ένα πλοίο τι γίνεται, εξετάσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρχουν οι συνθήκες οι κατάλληλε σε κάθε λιμάνι που να είναι ομοιογενεί στα διάφορα λιμάνια τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Υπάρχει αυτή η ιδέα τη ενία στηρίδα στα λιμάνια, αυτό πρέπει να αποτελέσει μια προτεραιότητα, μια... κάτι ουσιαστικό που θα πρέπει να αναφερθεί. Δεν θέλουμε μόνο απλούστευση των διαφόρων εντύπων, των διαδικασιών αυτών, αλλά χρειάζεται και μια απλούστευση όσον αφορά τις φυσικές υπηρεσίες που παρέχονται στα πλοία. Ίσως ε, είναι και θέμα οργάνωσης των λιμάνιων, θέμα χωροταξίας των λιμάνιων πρέπει να εξεταστεί και να ληφθεί υπόψη. Ίσως θα ήταν καλύτερο να γίνει μια κρόαση και στην Επιτροπή μας να ακούσουμε και τις αρχές τις λιμενικές φορείς που άμεσα έχουν ρόλο να διαδραματίσουν όσον αφορά τη διοργάνωση των αστηριοτήτων στα λιμάνια. Δεύτερη πρόταση. το ρόλο να είμαι ξεκάθαρος. Λοιπόν, ας πούμε ότι απλουστεύουμε και σε μερικά χρόνια έχουμε αποφασίσει ότι χρειάζονται κάποιες προδιαγραφές. Και ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφέ στην Ευρώπη που εγγυώνται μια ισορροπία και ομοιογένεια που προωθεί την ανταγωνιστικότητα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, θεωρούμε, υποθέτουμε. Διαφάνεια, ε, όσον αφορά τι υπηρεσίε, έχουν προσθεθεί διαδικασίε κλπ. Αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα την επόμενη μέρα τι θα κάνουμε. Όταν αλλάξουμε τα ρούχα μα, α πούμε, αλλάζουμε τα ρούχα που παρουσιάζουμε, την εικόνα που παρουσιάζουμε προ τα έξω, στον IMO. Το πώ λειτουργεί η Ευρώπη δηλαδή. Όσον αφορά όμω τι δράσει στα διεθνή ύδατα, θα πρέπει να έχουμε σωστή προσέγγιση. Η απλούστευσή μας να προβλέπει μελλοντικέ εξελίξεις στο διεθνέ προσκήνιο. Σταματάω εδώ, Πρόεδρε. Θα ευχαριστήσω εκ νέου τον εισηγητή και περιμένω να ακούσω τι θα πει σήμερα η Επιτροπή σας, τι απόψει θα ακούσουν στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ κύριο Μπεσέ από τους Πράσινους. Σας ευχαριστώ κύριε. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να πω εκ μέρους των Πρασίνων ότι εμείς θα υποστηρίξουμε οτιδήποτε πηγαίνει προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης ε, της ε, ε, θαλάσσιας κυκλοφορίας, της ροής της, της καλής ροής της και της αποτελεσματικότητάς της. τις εναλλακτικές ε, στις οδικές μεταφορές ε, αγαθών. Αυτή η βελτίωση, ο έξω ορθολογισμός των διαδικασιών, αυτή η εναρμόνιση των τεχνολογιών ε, της πληροφορίας μας ενδιαφέρει πολύ παρά το γεγονός ότι εσείς κύριε Στέρξ αναφέρατε και κάποια σημαντικά προβλήματα θα υπάρχουν δεν μας φαίνεται όμως ότι αυτά είναι ανυπέρβλητα εμπόδια για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας, ε, της, ε, τους, ε, τις ώρες διέλευσης κλπ. βεβαίως ε, να πούμε από την ε, γραφειοκρατία ε, όπως είπε ο προλαλής σας συνάδελφος, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι παναχωρούμε ως προς τις διαδικασίες ελέγχου. Η απλοποίηση δεν σημαίνει και απορρίθμιση. Και αυτό θα θέλαμε να το τονίσουμε. Πίσω από τις νέες τεχνολογικές προόδους και την εναρμόνιση ε, δεν εξαφανίζονται τα εμπόδια όσον αφορά την ασφάλεια ε, στις θαλάσσιες οδούς και την προστασία του περιβάλλοντος ε, επί των ζητημάτων αυτών. Λοιπόν, θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πλαίσιο της νέας αυτής οδηγίας. Υποστηρίζουμε βέβαια το στόχο της και θα προσπαθήσουμε να μην παρεκκλίνει από την βασική της πορεία. Ευχαριστώ. Thank for the ECR, Mrs. Foster. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στέρξ, όπως πάντα παρουσιάζει πολύ καλά τα πράγματα και αυτό που θέλει να πει και την άποψή του και κλείνει το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Εντάξει. Ναι, έλεγα ευχαριστώ στον κύριο Στέρξ, γιατί πιστεύω ότι είναι ο σωστός άνθρωπος ε, στη σωστή θέση. Έχει πάρα, πολύ γνω, πολλές γνώσεις στον τομέα και νομίζω ότι παρουσιάζει τα επιχειρήματά του πολύ σωστά, όπως είπα. Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που ετέθησαν ήδη είναι η λύση για τέτοιου είδου προβλήματα. Δηλαδή, φεύγει κάποιο από κάπου και ο στόχος είναι να φτάσει κάπου ε, με έναν τρόπο αρκετά απλοποιημένο, να μην υπάρχει πάρα πολύ και βαριά γραφειοκρατία και να μην ε, ξεκινάει από κάποιο από κάπου που είναι όλα τα πράγματα πολύ καλά και μετά καταλήγει κάπου που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν εξετάζουμε ένα τέτοιο θέμα και θα ήθελα να το τονίσω. Τώρα, Κάτι ακόμη για το οποίο η Επιτροπή μπορεί να μου απαντήσει. Υπήρξαν κάποια ζητήματα στις πρώτες συζητήσεις που κάναμε με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα επηρεάσει τις ε, χερσαίες περιοχές, σε περιοχές που δεν έχουν ε, ε, πρόσβαση στη θάλασσα, για παράδειγμα αν κάποιος είναι στο Λουξεμβούργο, και πώς θα συμπεριληφθούν οι συγκεκριμένες χώρες Κάτι ακόμα, ε, κάποιες άλλες ανησυχίες που εκφράστηκαν από κράτη-μέλη στο Συμβούλιο όσον αφορά τη σχέση με άλλα ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα, όπως για παράδειγμα η Σέγγεν, ε, ε, συστήματα παρακολούθησης σκαφών κλπ. Αν λοιπόν ε, προχωρήσει το θέμα, αυτά είναι ζητήματα που πρέπει οπωσδήποτε να τεθούν στην αρχή της διαδικασίας, ε, ώστε να γνωρίζουμε τι γίνεται. Κύριε Στέρξ, ίσως να μπορείτε να μου απαντήσετε. Όσον αφορά την προθεσμία, νομίζω ότι θα δούμε, να σας πω την αλήθεια, πώς θα πάνε τα πράγματα. Και όσον αφορά τη, τη διατύπωση, ε, τη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουμε, Όχι ότι ως Αγγλίδα είμαι προκατηλημένη, αλλά νομίζω ότι όταν μιλούμε για διεθνείς μεταφορές πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο περίπλοκα τα πράγματα ε, και μιλάω για τη χρήση της αγγλικής γλώσσας. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο απλά και αυτό ίσω να είναι υπέρ τη χρήση αγγλική γλώσσα. Διαφορετικά θα υπάρχει πολύ μεγάλη σύγχυση. Ε, βέβαια υπάρχει και το θέμα των γλωσσών ε, που πολλοί δεν έχουν όταν φτάνουν σε ένα συγκεκριμένο λιμάνι. Και είναι ένα ζήτημα αυτό. Για τα υπόλοιπα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Στέρξ για την παρουσίασή του και είμαι βέβαιη ότι τα πράγματα θα ε, συνεχίσουν όπως πρέπει. Ο κύριος Βαντάλεν. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Στέρξ είναι ο εισηγητής για το θέμα αυτό. Γιατί συμπεριλαμβάνεται το Στέρξ το όνομά του που σημαίνει ισχυρός στα Ολλανδικά. Οπότε Έχουμε το θέμα των διατυπώσεων και έχουμε και το θέμα της ε, γραφειοκρατίας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μιλήσατε για την ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό να ξέρει κανείς και τι εμπόρευμα ε, έχει ένα πλοίο όταν πρόκειται να ε, εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ προσφάτως διερεύνησα τα ατυχήματα στη θάλασσα και πολλές φορές δεν γνωρίζαμε καν τι εμπόρευμα έχει το πλοίο. Πώς είναι δυνατόν να ανταλλάσσει πληροφορίες αν δεν γνωρίζεις ακριβώς τι κουβαλάει το πλοίο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και θα ήθελα να μου πει και η Επιτροπή ποια είναι η άποψή της. Δεύτερο θέμα που θα ήθελα να θέσω, κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στο τι συμβαίνει στην πράξη και το τι συμβαίνει στο χαρτί. Πώς γίνεται λοιπόν η πρόσβαση στις πληροφορίες, αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει επίσης να ορίσουμε το δικαίωμα της πρόσβασης στα δικαιώματα της πρόσβασης. Ποιος θα έχει τα δικαιώματα αυτά. Πάρα πολλές ήταν οι πληροφορίες που υπάρχουν και επίσης υπάρχει και το ζήτημα του, όπως είπα, της πρόσβασης στα δικαιώματα και συμφωνώ με τον συνάδελφο από τους πράσινους. Πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός. Ποιος έχει πρόσβαση σε τι. Και επίσης ε, υπάρχει και το πρόβλημα της εποπτείας της όλης διαδικασίας. Όσον αφορά τη γλώσσα, κοιτάξτε. Εμένα μου φαίνεται πολύ σημαντικό να μπορεί ο καθένα να μιλάει τη γλώσσα του. Αλλά εν προκειμένου θα ήμουν υπέρμαχο τη χρήση της αγγλικής γλώσσας. Γιατί, καταλαβαίνετε, διεθνεί μεταφορές, διαθαλάσσεις για παράδειγμα, Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι ναυτικοί ε, καταλαβαίνουν κάποιο είδους αγγλικά, οπότε πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε την αγγλική γλώσσα ως γλώσσα επικοινωνία Αυτό βέβαια πρέπει να συνδεθεί και με άλλου τομεί μεταφορών ε, ενδεχομένως. Για παράδειγμα, οδικές μεταφορές και ε, εσωτερικές ε, μεταφορές των ε, εσωτερικών οδών. Οι περισσότεροι ναυτικοί μάλιστα προέρχονται από γλώσσες αγγλόφωνες, Φιλιππίνες για παράδειγμα. Και εν πάση περιπτώσει ήθελα να πω ότι η αγγλική γλώσσα όλο και περισσότερο χρησιμοποιείται στις ε, ε, ε θαλάσσιες μεταφορές και γενικότερα εν πλώ, οπότε εν προκειμένου μπορώ να υποστηρίξω τη χρήση της αγγλικής γλώσσας. Τώρα, ένα ερώτημα ή ο εισηγητή θα μου απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορά το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Μιλάμε για μεταφορές ε, μικρών αποστάσεων, αλλά δεν αναφέρεται πουθενά αυτός ο όρος στο άρθρο 2. Εδώ λέει ότι μιλάμε για πλοία που φεύγουν και φτάνουν σε κοινοτικά λιμάνια. δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένες μεταφορές ε, μικρών αποστάσεων ή όχι. Πρέπει να γίνει μία διάκριση γιατί είναι γενικόλογη κάπως η ε, διατύπωση. Πρέπει να κάνουμε μία γενικολογικα λογικα μεταξύ μεγαλύτερων αποστάσεων, μεταφορών μεγαλύτερων αποστάσεων και μικρότερων. Και αν δει κανείς την πρόταση, δεν, αναφέρεται καθόλου η, ε, δεν ε, αναφέρονται καθόλου μεταφορές μικρών αποστάσεων. Πριν απαντήσει ο κύριος Τίλμαν, λέει ο πρόεδρος, ε, όσον αφορά τις ε, χώρες που δεν έχουν θάλασσα.